που έχει τα σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδίω στι Βρυξέλλε. Τίποτα άλλο και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δία Μέρα. Έχει κλείσει η συζήτηση λοιπόν και θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή αύριο αν θέλει ο Θεός βέβαια. Ακολουθεί η σειρά των μονόλεπτων ομιλιών. Βάσει το άρθρο 150 του κανονισμού. Δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Τισέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τώρα εξετάζει την συνολική συμφωνία μπανάνας ε, που επιτεύχθη στα ΟΜΠΟΕ ε, και το σώμα θα κληθεί να αποφανθεί για τους δασμούς, εισαγωγικούς δασμούς για την μπανάνα, για ε, τις αγωγές από τη Λατινική Αμερική. Οι υπερπεριφερειακές ε, ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Μαδέρα ή τα Κανάρια νησιά που πλήττονται θα χάσουν πάρα πολλά από αυτή την συμφωνία και Εάν πρέπει να απαιτήσουμε από τους άλλους ε, τις ίδιες απαιτήσεις ε, για την υγιεινή παραδείγματο χάρη, ε, τις συνθήκες εργασίας ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο δίκαιο και πρέπει να υπάρχει και ένα αντιστάθισμα για τις απώλειες που θα υποστούν ε, οι παραγωγοί σε αυτές τις υπερπεριφερειακές ζώνες της Ένωσης. θα πρέπει να βρουν κάποια άλλη απασχόληση, διότι όπως έχουν τώρα τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν με αυτή την δραστηριότητα. Στις συμφωνίες υπάρχουν οι νικητές και οι τιμένοι και θα πρέπει να φροντίσουμε τους ιτημένους. Ευχαριστούμε κυρία Μπρινκέβιτσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη ο αριθμός των ατόμων που η μόνη πηγή εισοδήματός τους είναι η σύνταξή τους αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα. Άνθρωποι που εργάστηκαν σκληρά όλη τη ζωή, που μεγάλωσαν τα παιδιά τους, πλήρωσαν φόρους, έκαναν περαίωση στις χώρες τους, περιμένουν να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι σαφές μέσα στην οικονομική κρίση. Όταν αυξήθηκε η κρίση δεν ακολούθησαν οι, οι συντάξεις πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βοηθούν και τα άνεργα παιδιά τους. Στη Λιθουανία μειώθηκαν οι συντάξεις και τα άλλα επιδόματα. Σήμερα γίνονται πολλές συζητήσεις για την πρόταση της Κομισιόν να αυξηθεί η ηλικία σύνταξης. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει καμία λύση για την απασχόληση των ηλικιωμένων. Εκατομμύρια ατόμων μπορούν να παγιδευτούν στην ε, ένδια σε μια ηλικία πριν από την σύνταξη όσο γίνεται και πιο μακρινή η, προ... η προοπτική της σύνταξης. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό ότι βάζουμε ανθρώπους σε μια ευάλωτη κατάσταση γιατί έχουν μερική απασχόληση, δεν έχουν ε, υποστήριξη λόγω άδεια μητρότητα κτλ. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να βρουν άλλες λύσεις για να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή για τα άτομα σε ηλικία ε, σύνταξη. Κυρία Μουσμπένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σήμερα έχουμε δύο επέτειους, ε, την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία. Επίσης, είναι η μέρα της ελευθερίας έκφρασης στη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Μην ξεχνάτε το πολιταρχικό καθεστώς, μην ξεχνάτε την ε, ε, τρομοκρατία που ε, δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο και δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία φαίνεται χωρίς να παραβιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, χωρίς να παραβιάσουμε την ελευθεροτυπία. Εάν χρησιμοποιήσουμε περιφερειακέ οργανώσει, αν δεν φτιάξουμε ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για γρήγορη ε, προειδοποίηση, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κορομέβα ή Ρουέδε. Είχα προειδοποίησει ότι θα γίνει αυτό στην προηγούμενη Ολομέλεια και έγινε πια. Αυτή τη στιγμή ο λαό των Σαχαραουί θρυνεί 19 νεκρούς και ε, πάνω από 700 εξαφανισμένους. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες των χωρών μας λένε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και δεν πρέπει να, επα... να επέμβουμε, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια στο Μαρόκο. Όχι κυρία Άστον, όχι κύριε Χιμένες, όχι κύριε Κουσνέρ. Τα θέματα των φόνων και των εξαφανίσεων είναι πολύ απλά θέματα. Η θέση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί αυτών είναι πολύ απλή και αυτή θα πρέπει να ζητήσουμε ευθύνε από την κυβέρνηση του Μαρόκου και να απορρίψουμε τη στάση του. Μέχρι να γίνεται αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε το διμερές εμπόριο για το Μαρόκο και τα προνόμια που απολαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει αυτό το εμπόριο που γίνεται σε βάρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Ο κ. Μιγάλσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δηλώσω πολύ χαρούμενος που ε, είναι εδώ ακόμη η Επίτροπος διότι ε, θα την ενδιαφέρει το ζήτημα. Δεν πρόκειται για αστείο. Ε, από τις 4 μέχρι 6 Οκτωβρίου ένας δημοσιογράφος ε, στη Ρωσία ε, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μπροστά στο σπίτι του. Σίγουρα το έχετε ακούσει. του έσπασαν το πόδι, τα δάχτυλα και πήγε στο νοσοκομείο. Δεν είναι η πρώτη τέτοια επίθεση που γίνεται σε δημοσιογράφους στα, πέρα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Πολωνοί που εμπειρογνώμονες για τα θέματα της Ρωσίας δήλωσαν ότι 300 δημοσιογράφοι απεβίωσαν ε, πέρυσι στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το αναφέρω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, ο σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων. Όταν συζητάτε λοιπόν με του ε, συναδέλφου σα, υπενθυμίστε του ότι πρέπει να παρεμποδίσουμε τέτοια συμβάτα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τέτοιο διάλογο, εν τη αυτή περιπτώσει ο κύριο Φερέιρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στην πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που ισχύει στην Δυτική Σαχάρα. Η Σαχαρουή έχουν ε, κάνει μια ενέργεια διαματηρίας για τις συνθήκες ε, διαβίωσης τους καταβλισμούς τους <clears throat> και θέλουν να εξασφαλίσουν το δικαίωμά τους για την αυτοδιάθεση. Η καταστολή από την αστυνομία της, ε, του Μαρόκου <clears throat> οδήγησε σε καταστροφή αυτόν τον καταβλισμό και οδήγησε σε εκατοντάδες ατόμων που εξαφανίστηκαν και δυστυχώς δεκάδες νεκρών. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην αποστροφή μας ως Ευρωπαίων, γιατί και εξάλλου πολλοί από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απελάθηκαν από τις ε, αρχές του Μαρόκου και δεν επέτρεψαν σε αυτούς να πλησιάσουν. Επίσης και ένας βουλευτής από το κοινοβούλιο μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Νεολαίας σε παγκόσμιο επίπεδο και πολλοί δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν και αυτοί να πλησιάσουν την Δυτική Σαχάρα. Θα πρέπει να κρούσουμε τον κόνδυνα του κινδύνου ότι είναι ε, επονίδη της στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την τύχη τόσα χαρούι και η υποστήριξή τους προς μια χώρα που φέρεται με τέτοιο τρόπο και απολαμβάνει τόσα προνόμια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέζιο είναι ακόμα επόμενος Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ευστήσω την προσοχή όλων και κυρίως του Προέδρου του Κοινοβουλίου ε, σε μία απόφαση που εξεδοθεί πρόσφατα για την εντολή της Επιτρόπου και να σας χαιρετήσω κιόλας, δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα. Ε, και η απόφαση φέρει επί το πεδίο εφαρμογής μιας πολύ σημαντικής οδηγίας ε, που σχετίζεται με την τρομοκρατία. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την προσέγγιση για την προστασία των πολιτών που θέλουν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την υποβολή αίτησης ασύλου ή με το να θεωρηθούν ως πρόσφυγες. Αυτή η τελευταία ε, απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τους δίνει τη δυνατότητα προστασίας ενώ δεν την αξίζουν. Εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι λόγω τρομοκρατίας σημαίνονται στην Ευρώπη. Ε, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει, να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση αυτή της οδηγίας, ώστε αυτέ οι παρερμηνίε του δικαίου να αποφευχθούν. Thank you, Mr. President. Last Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μετακίνηση στο Στρασβούργο θα αποτελέσει αύξηση των δαπανών μας κατά 5,9% του προπολογισμού. Είμαστε μέσα σε μια οικονομική κρίση και τα θύματα στη δική μου εκλογική περιφέρεια, στα West Midlands δηλαδή, διαμαρτύρονται οι φοιτητέ θα πληγούν ιδιαίτερα από τα μέτρα λιτότητας γιατί αυξάνονται κατά το τριπλάσιο σχεδόν τα δίδακτρα. Το... Οι αυριανές δεξιότητες των ανθρώπων θα βασίζονται στους νέους. Αυτούς πρέπει να προσέξουμε και προειδο... σας προειδοποιώ όλο και περισσότεροι θα διαδηλώνουν και θα διαμαρτύρονται. Κυρίες και κύριοι, πιέστε ήρεμοι τη σαμπάνια σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν θα σας αφήσουν ήσυχους. Η κυρία Βασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην διάσκεψη κορυφής του Δουνάβη της 8 ε, ε, Νοεμβρίου ήταν παρούσα Παρούσε αντιπροσωπείε 14 κρατών που αντιμετώπιζαν την κατάσταση του Δούναβη. Ήταν επίση και η Δημοκρατία τη Μολδαβία, που είχε και μια περαιτέρω ευκαιρία να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πολύ πρόσφορη στιγμή, διότι στο τέλο του έτου θα εγκριθούν τα βασικά έγγραφα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του Δούναβη και το, 12, το 2011 θα αρχίσει η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Ήταν πολύ σημαντική λοιπόν η συμμετοχή του κ. Μπαρόσο και, του, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια χρηματοδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ και με ότι με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσουμε και περαιτέρω πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την περιοχή του Δούναβη. Η Ευρωπαϊκή Στατική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δούναβη έχει υποστηριχθεί από το 2008 από την Ρουμανία, η αέναε λοιπόν εφαρμογή αυτών των μέτρων θα επιτρέψει και την οικονομική ανάπτυξη των νότιων περιοχών της Ρουμανίας. Ευχαριστώ και Μουλτσουμέσκ. Η κυρία Μουνίθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των Ισπανών Σοσιαλιστών θέλω να εκφράσω την ε, βαθιά μας ανησυχία για τη βία στην ε, ε, Δυτική Σαχάρα και το Μαρόκο. Εκφράζουμε λοιπόν τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα οποία έγιναν εκεί. Είναι συγκεχημένες οι ειδήσει που ήρθαν από εκεί και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή έρευνα και να έχουμε διαφάνεια στα επίπεδα της επικοινωνίας. Είναι μεγάλη σημαντική η στρατηγική σημασία του Μαρόκου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσθέσει, να προσθέσει και τη δική της φωνή στις διεθνείς δυνάμεις που ζητούν να υπάρξει διάλογος. <clears throat> και η Ισπανία το υποστηρίζει. Παρά λοιπόν τη σοβαρότητα των ε, γεγονότων είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών και να παραμείνουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη έχει ιστορία πάνω από 30 ετών και θα πρέπει να καταλήξει με μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στα πλαίσια του, <clears throat> του ΟΗΕ ώστε μεταξύ του Μαρόκου και του λαού του Σαχαραουή να μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος έχει υπερασπιστεί τα πολιτικά δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτό και εξεπλάγει όταν έμαθα στην προηγούμενη σύνοδο το Κοινοβούλιο τελικά δεν τοποθετήθηκε για τις ε, τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές ε, στην Ουκρανία παρά τις αξιόπιστες ε, και εξαιρετικά ανησυχητικές πληροφορίες που είχαμε για την παρενόχληση δημοσιογράφων, μελών της αντιπολίτευσης από τους εκπροσώπους του κυβερνώντος κόμματος σε διάφορες περιφέρειες Ουκρανίας. Ανεβλήθησαν οι εκλογές και ε, μάλλον, συγγνώμη, αναβλήθηκε η απόφαση του, περί του ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, δι... Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί η Κομισιόν εχθές επιβεβαίωσε μια στρατηγική 2021 που στηρίζει τη διεύρυνση προς τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και γιατί είχε αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίξει τις χώρες αυτές στην ενταξιακή τους πορεία. Χαίρομαι επίσης για την έγκριση μέτρων όπως την κατάργηση των θεωρήσεων για τις χώρες αυτές, για, όπως για το Μαυροβούνιο που έχει αυτή τη στιγμή καθεστώς υποψήφιας χώρας. Επίσης σημειώθηκε πρόοδος στι διαπραγματεύσεις με την Σερβία Παρ' όλα αυτά παραμένουν ορισμένα προβλήματα όπως η σύναψη διαλόγου μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή αυτή και διαπραγματεύσεις για το όνομα της Μακεδονίας. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση προς την Βοσνία Ερζεγοβίνη και να αρχίσει η διαδικασία απελευθέρωση των θεωρήσεων και για το Κωσυφοπέδιο. Για όλα αυτά χρειάζεται σαφή στρατηγική και όραμα ώστε να πλησιάσουν πράγματι οι χώρες αυτές περισσότερο προς την Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούκαν. Και τώρα ο κύριος Μιλάνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, επί σειρά ετών το Μαρόκο αρνιόταν ότι ήταν σε πόλεμο, σε, πολεμική σύραξη με τους Σαχράουι. Ε, σήμερα υπάρχει ε, υπερβολική καταστολή αυτών των ανθρώπων που το μόνο που κάνουν είναι να διεκδικούν το δικαίωμά τους να ζουν ελεύθερα. Ε, το Μαρόκο επεξέτεινε αυθαίρετα τα σύνορά του ε, εμείς ε, δεν μπορούμε καν να μεταβούμε ε, επί επιτόπου για να διαπιστώσουμε τι γίνεται ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ε, παραπέμπει στη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ. Εδώ και 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνει ε, και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Οπότε ένα μήνυμα προς την κυρία Άστον και προς το Κοινοβούλιο. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει ε, να διακόψουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τις εμπορικές συμφωνίες παραδείγματος χάρη και να μην ανανεώσουμε τις αλληλευτικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε κύριος Λούχαν. Zilele acestea au fost aduse în prim plan. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πρόσφατα ε, τονίστηκαν στη συζήτηση πολλά στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομία. Ε, τώρα νομίζω ότι χάρη στα νέα μέτρα θα μπορέσει η Ένωση να δράσει επί τη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ε, βασική η πρωτοβουλία, αλλά μην ξεχνάτε για την ε, επόμενη πενταετή περίοδο προγραμματισμού η συζήτηση και ο διάλογος θα πρέπει να ξεκινήσει σε περιφερειακό επίπεδο, ούτω ώστε να ε, ξεκινήσουν πραγματικά και όλες οι υπόλοιπες διασυνοριακές, διαπεριφερειακές δράσεις. Για την επόμενη περίοδο κάθε περιφέρεια θα πρέπει να τοποθετηθεί και να δράσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι διαφορετικοί φορείς ώστε να εντοπίσουμε το δυνατό σημείο κάθε περιφέρειας και το σωστό χρονισμό για να δράσει, για να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της. Ε, απευθύνω έκκληση στις περιφέρειες να συμμετάσχουν στις εταιρικές ε, σχέσεις στο δικό τους επίπεδο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καστίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ΓΑΜΑ 20 αρχίζει στη Σεούλ και από μεταξύ των θεμάτων του θα είναι και η οι εισαγωγές σπανίων πρώτων υλών από την Κίνα που χρησιμοποιούνται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είναι θέμα νέων τεχνολογιών και επιστημονικής έρευνας και μπορεί η μείωση των εξαγών αυτών να απειλήσει το μέλλον της Ευρώπης είναι απαράδεκτο το μέτρο αυτό που έλαβε η Κίνα και ζητώ του προσώπους της Ένωσης μαζί με τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες χώρες όπως την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στο γάμα 20 και να καταδικάσουν την αυθαίρετη αυτή πράξη της Κίνας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τσουκάου. Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γυράσκει και λόγω της οικονομικής κρίσης έχει φτάσει το 10% ο αριθμός των ηλικιωμένων. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε βιώσιμα συστήματα συνταξιοδότησης. Διότι πρέπει να υπάρξει μία εγγύηση ενός κατωτάτου εισοδήματος για μία αξιοπρεπή ζωή. Το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού αυξάνει, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να αυξηθεί το όριο της συνταξιοδότησης. Μπορεί μεν να είναι ικανοί και οι γυρεότεροι να συμβάλλουν στην οικονομική ζωή, αλλά δεν πρέπει να υποχρεώνονται σε αυτό. Ε, τη στιγμή μάλιστα που άνθρωποι που καταφανώς είναι σε κατάσταση όπου είναι ικανοί να εργαστούν δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας. Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης λοιπόν οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεργία. Ευχαριστούμε κύριε Μικουλάσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σήμανση των τροφίμων είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερος τους πολίτες της Ένωσης. Έχω καλά νέα. Από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου οι πολίτες της Σλοβακία δεν ενδιαφέρθηκαν μόνο για την πρώτη ανάγνωση της συμφωνίας για την έκθεση Σόμερ αλλά ε, Η βιομηχανία τροφίμων, το πανεπιστήμια ενεπλάκησαν, ε, νέοι συμμετείχαν στις ε, συζητήσεις. πήρεξε μεγάλη κινητοποίηση. Και, ο Γερμαν... και η Ρενάτα Σόμερη, η Γερμανίδα συνάδελφός μας, ενεργά μετήχε μαζί με άλλους τρεις βουλευτές από τη Σλοβακία ε, και ε, αυτό δείχνει πόσο μπορούν να καταφέρουν ε, σε μια συμμετοχική δημοκρατία οι βουλευτές. Έτσι μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστούμε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πρατισλάβα. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην περίπτωση της ε, Σνικιάνη, η οποία στο Ιράν επρόκειτο να ε, θανατωθεί δια, λιθοβολισμού δια υποτιθέμενη ε, μοιχεία. Αλλά χάρη στην διεθνή πίεση έχει μετατραπεί σε ισόβια Τώρα με αποχωρισμό και όχι με λιθοβολισμό. Ε, υπήρξαν 270 αιτήσει ε, ε, στο διαδίκτυο και επίσης η παρέμβαση του πρόεδρου Σαρκόζη ο οποίος έκανε και μια προσωπική παρέμβαση έτσι έχει ε, αναβληθεί η εκτέλεση θανατικής ποινής που επρόκειτο να γίνει στις 3 Νοεμβρίου. Αλλά υπάρχει η πρόθεση της Ιρανικής κυβέρνησης να εκτελέσει τις ακίνες. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει όλες τις προσπάθειες για να μπορέσει να απελευθερωθεί και να σταματήσει ο κρατικός φόνος γυναικών και άλλων ε, ανθρώπων που θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής στον γύρο αυτό ομιλιών ενός λεπτού. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Θωμά Μαν για τη δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη